Τελευταία ήταν αυτή η παρατήρηση που είχα να κάνω για να ξέρουμε τι συζητάμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ στον Πολύ Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Η ψηφορία θα γίνει αύριο. με τη ημερησία διάταξη. Έκθεση Μπελέτ. Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα να δινέσει στα τρόφιμα και τι ζωοτροφέ. 0001 2011. Θα να δώσω το λόγο στον εισηγητή καταρχήν για τέσσερα λεπτά. Well, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Ε, συζητούμε εδώ για τα υγιεινά ε, τρόφιμα και ζωοτροφές. Ε, είναι κέρια σημασία ε, το ζήτημα. Θα συμφωνήσετε. Ε, σε καμία περίπτωση δεν ε, πρέπει να ε, επιτρέψουμε να υπάρχει φυσικά ραδιενεργός ακτινοβολία, αλλά χρειαζόμαστε ένα κανονισμό για περιπτώσεις ανάγκης. Υπάρχει εδώ και 20 χρόνια αυτός ο κανονισμός και πρέπει να επικαιροποιηθεί, γιατί έχουν σημειωθεί άλλες εξελίξεις. Ελπίζω, έχουν γίνει αλλαγές λοιπόν στον κανονισμό που βελτιώνουν τον κανονισμό και ελπίζω ότι θα τις εγκρίνεται στην αυριανή ψηφοφορία. Ε, ελπίζω να με ακούει ο Επίτροπος, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είναι ε, απαραίτητο να μπορεί σε επίγουσες καταστάσεις ε, η Επιτροπή και όχι το Συμβούλιο ε, να ασκεί τις εκτελεστικές εξουσίες. Μετά από ένα ατύχημα πυρηνικό η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την ηγετική ε, θέση στις ε, προσπάθειες. Ε, μετά το Τσέρνομπιλ συστήθηκε το σημερινό σύστημα, το 85 δηλαδή, και έχουν σημειωθεί εξελίξεις, έχει τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και άρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε και τον κανονισμό. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει διόντως υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες τεχνικές προδιαγραφές. Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγιεινής, των τροφίμων και της δημόσιας υγείας έχουν γνωμοδοτήσει και εξυπακούεται παρότι δεν προβλέπεται ε, στον ισχύοντα κανονισμό. Προκύπτει λοιπόν με σαφήνεια ότι οφείλουμε να επικαιροποιήσουμε τα επιστημονικά δεδομένα του κανονισμού. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου να μας υποβάλει έκθεση για την προσαρμογή των τεχνικών προτύπων προτύπων και προδιαγραφών ε, και αν χρειαστεί να εμβαθύνεται αυτή την, ε, ίσονος, ε, αυτόν τον ίσονο σημασίας κατάλογο όπως ονομάζεται για τα τρόφιμα. τρίτη παρατήρηση, Πρόεδρε, ο ορισμός της βρεφικής τροφής. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα και ε, χρειαζόμαστε ε, προσαρμογή του κανονισμού γιατί ισχύουν πλέον νέα δεδομένα, νέες νομικές πράξεις ε, για την προστασία αυτών των τροφίμων. Αυτό θα το ζητήσουμε αύριο και στην Ολομέλεια. Ε, τέταρτον, προτείνει το Κοινοβούλιο ε, να ε, αποζημίωση για τους γεωργούς που πλήττονται από τέτοιου είδους πυρηνικά ατυχήματα. Δεν προβλέπεται αυτό, αλλά θα θέλαμε, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια σχετική πρόταση. Τέλος, το θέμα της νομικής βάσης. Πρόεδρε, με ομοφωνία η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του ε, Κοινοβουλίου γνωμοδότησε ότι το άρθρο 168 εδάφιο 4 της συνθήκης πρέπει να αποτελέσει τη νομική βάση αυτής της πρότασης και σας παραθέτω το σχετικό τμήμα της ε, συνθήκης. Ε, πρόκειται για τα που επηρεάζουν άμεσα την δημόσια υγεία. Τέλος παράθεσης, ε, σίγουρα είναι σημαντική η αλλαγή γιατί θα χρησιμοποιηθεί μάλλον συναπόφαση, δηλαδή είναι συνήθινη νομοθετική διαδικασία σε σχέση με τον τωρινό κανονισμό που συνδέεται ακόμη με τη συνθήκη Ευρατών. Ε, νομίζω ότι είναι προ συμφέρον όλων των Ευρωπαίων αύριο να εγκριθεί η πρόταση για την αναδιατύπωση του κανονισμού. Σα ευχαριστούμε εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να συγχωρέσετε τον κύριο Σέρκοβιτς και Ότιγκερ που μου ζήτησαν να τους εκπροσωπήσω γιατί έχουν άλλες ε, δεσμεύσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή σας γιατί που τόνισε όλες τις πτυχές ενίσχυσης ε, της, ε, της προστασίας των τροφίμων και των ζωοτροφών από τη ραδιενέργεια. Ξέρετε ότι ο 3954 του 87 του Συμβουλίου αναφέρεται στο προήμιο λέγοντας ότι μόνο το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για αυτού του είδους της ρυθμίσεις. Όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να δεχθεί όλες τις τροπολογίες της έκθεσης Μπελέτ. Ο πρώτος ε, λόγος αφορά στην συμφωνία, στη διαθεσμική συμφωνία επανίδρυσης των τριών θεσμικών οργάνων όπου τα κωδικοποιημένα μέρη δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και αυτό για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την συνοχή όλων των μέτρων ο σεβασμός αυτής της συνενετικής διαδικασίας είναι σημαντικός για να διατηρηθεί η διαθεσμική ισορροπία και το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Κομισιόν. Το σπάσιμο αυτής της ισορροπίας θα καθιστούσε de facto ανεφάρμοστη αυτή την νομοθετική διαδικασία. Και αυτή η νομοθετική διαδικασία όμως έχει ως στόχο το να νομοθετούμε καλύτερα ενισχύοντας τη διαφάνεια στην υπηρεσία των πολιτών. Δεύτερος λόγος αφορά στην ουσία. Η πρώτη τροπολογία που ψήφισε η Ήτρε αφορά στη νομική βάση. Η συνθήκη 31 της ΕΡΟΑΤΟΜ θα αντικαθιστιόταν από το άρθρο 168 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες τροπολογίες συνδέονται με αυτή την αλλαγή της νομικής βάσης. Θεωρεί η Κομισιόν ότι η τροπολογία για τη νομική βάση είναι αδικαιολόγητη. Είναι και αντίθετη με το άρθρο 106α της συνθήκης Ευρατόμ που λέει ότι όταν υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για ένα ειδικό θέμα η συνθήκη Ερατόμ υπερισχύει της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε η εγκυρότητα του άρθρου 31 της συνθήκης ΕΡΑΤΟΜ έχει επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφαση σε 70 Τώρα για το κεφάλαιο 3 σχετικά με τις, ε, τις ακτινοβολίες ορίζονται οι κανόνες από την από το άρθρο 31 της συνθήκης Ευρατόμ. Αυτά είναι τα νομοθετικά όρια κύριε Πρόεδρε και βάσει αυτών των νομοθετικών ορίων η Κομισιόν θέλει να απορριφθούν οι τροπολογίες της έκθεσης Μπελέτ. Και αυτά εξ ονόματος του κυρίου Σέσκοβιτς και του κυρίου Όπλιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πίτρα Μπένια. Εξ στο των πολιτικών τώρα, δύο λεπτά εξ ονόμου του ΕΛΚ, η συνάδελφο Ιωντάν Σιζέλη. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Η ραδιενέργεια και η εκτενοβουλία είναι ε, ένα επικίνδυνο θέμα γιατί δεν, τη βλέπουμε, δεν την μυρίζουμε, δεν την ακούμε αλλά είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχει όμως και θετικά χαρακτηριστικά και αυτό χρησιμοποιείται και στην ιατρική και στην έρευνα για την δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις θετικές επιπτώσεις θα πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις για τους φόβους που έχουν οι πολίτες. Πρέπει να αυξήσουμε την ασφάλεια. Το έκανε πάρα πολύ καλά ο εισηγητής μας κ. Πελέτ προετοιμάζοντας τις τροπολογίες για τον κανονισμό που αφορά την μόλυση τροφίμων και ζωοτροφών σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Τον συγχαίρω και ελπίζω η Κομισιόν να αλλάξει τη θέση της και να λάβει υπόψη αυτά που προετοίμασε ο εισηγητής. Ελπίζω επίσης ότι το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη αυτά που έχει προετοιμάσει το Κοινοβούλιο και είμαι πολύ ε, απογοητευμένη που η εκπρόσωπος ε, του του Συμβουλίου δεν είναι πια παρούσα. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δεχθούν τις δημοκρατικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τότε που υιοθετήθηκε η συνθήκη Ευρωτόμ, το 58 δηλαδή, και να λάβουν περισσότερο υπόψη σε αυτά που αποφασίσαμε και υιοθετήσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις ακτινοβολίες και τις ιονίζουσες ε, ακτινοβολίες. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά ο κύριος Γκύρια Καζονάματος της ομάδας του. Πρόεδρε, το θέμα της παραγωγής ισοτόπων και των πειραματικών αντιδραστήρων για ιατρικούς και άλλους στόχους ε, είναι ένα θέμα που ε, απαιτεί την ε, ασφάλεια των προϊόντων, ασφαλείς τροφές, ασφαλή τρόφιμα. Πρέπει κάπως να μεριμνήσουμε για να τα εξασφαλίσουμε όταν σημειώνεται ένα τέτοιο ατύχημα. Οι βλάβες των πυρηνικών αντιδραστήρων ε, μας οδήγησαν στην έγκριση αυστηρών προτύπων για την προστασία από την ε, ακτινοβολία. Όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ε, σοβαρά όπως είχαν παρουσιαστεί. Υπήρχε μεγαλύτερη ραδιενέργεια, επιμόλυνση τροφών και τροφίμων από την ραδιενέργεια στις ευπαθείς περιοχές. Φαίνεται όμως ότι ήταν κάπως υπερβολική η αντίδραση και Τελικά επέστρεψαν οι άνθρωποι στα χωριά που είχαν εγκαταλείψει μετά ε, τα πυρηνικά μετά το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, παραδείγματος χάρη, και μάλιστα ισχυρίζονται ότι κάτω από ένα όριο μπορεί να είναι και ευεργετική ε, ε, η ακτινοβολία αυτή. Χρησιμοποιήθηκαν ε, και επιστημονικές ε, μελέτες ε, για να στοιχειοθετηθεί αυτό. Κατά μέσο όρο μπορούμε να απορροφήσουμε 2,7 μίλι το χρόνο και μετά από 70 χρόνια με τη συσσόρευση φτάνουμε στα 200. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε πραγματικά τις ραδιολογικές καταστάσεις ε, πήγουσας ανάγκης, να δούμε ποια είναι η ραδιενέργεια που προκύπτει από έκρηξη ηφαιστείου. του χάρη, οριζεται κάποιε τέτοιε περιπτώσει είναι πιο υψηλή η ραδιενέργεια παρά μετά από ατύχημα. Και πώς επηρεάζει το θηροειδή, του ιστούς, ε, τα οστά μας ε, και μετά τους επνεύμονες και, τα... και άλλα μέρη του σώματό μα. Η κυρία Χόλ. Νομίζω ότι είναι πολύ έγκαιρη η υποβολή τη πρότασης αυτής γιατί τον Απρίλιο φέτος θα έχουμε την 25η επέτειο από το δυστύχημα του Τσερνομπίλ. Θα θυμόσαστε πόσο ε, ανήσυχοι ήταν οι πολίτες τότε και πόσο υψηλά ήταν τα επίπεδα Μόλι σε ορισμένε ε, περιοχέ, όπω παραδείγματο χάνει στην περιοχή των λιμνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν οι κλαματολογικέ καταστάσει τέτοιε που η μόλυνση έμεινε πολλά χρόνια. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε τώρα ένα σύστημα που θα δώσει τι μεγαλύτερε διαβεβαιώσει στου πολίτε σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε διαφορετική νομική βάση. Η ομάδα των πυρογνωμόνων το διεύρυνε για να συμπεριληφθούν και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τα τρόφιμα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπορούμε να τα αφήσουμε στα χέρια των πυρηνικών εμπειρογνωμόνων. Είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό τα επίπεδα της επιτρεπόμενης ακτινοβολίας να είναι τέτοια ούτως ώστε τα τρόφιμα να μπορούν να καταναλωθούν από ανθρώπους κάθε ηλικία. Μπορούμε να φανταστούμε ποια προβλήματα θα υπάρχουν εάν παραδείγματος χάρη λεχθεί ότι τα καρότα φερρυπίν Μπορούν να το τρώνε οι ενήλικες αλλά όχι τα παιδιά. Χρειαζόμαστε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί ο καθένας να ε, έχει εμπιστοσύνη σε αυτές και θα ήθελα να είμαστε ο, όπως το, οι Ηνωμένες Πολιτείες και να ορίσουμε για καθένα το ανώτατο ετήσιο ε, ε, όριο σε ένα μακροσίλβερ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε παραδείγματος χάρη ε, τις ε, παραδόσεις ε, που υπάρχουν, η κασάδα παραδείγματο χάρη, είναι κάτι, ένα τρόφιμο βασικό για ορισμένους, όχι για όλους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Μπέλε για την πολύ συνεννητική στάση που ακολούθησε και ελπίζω η Κομισιόν να μην ξεχάσει ότι το Κοινοβούλιο είναι σημαντικά ενωμένο σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Πρώτα, σε ευχαριστώ κυρία Χολ. Επόμενη για δύο λεπτά εξ των Πρασίνων, η κυρία Χάρμς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, αυτές οι προτάσεις τη Κομισιόν μα απασχολούν γιατί η, ε, ο ισχύων κανονισμό ε, έληξε το 2010 και κατά την επεξεργασία της πρώτης αυτής θυμήθηκα όπως με την Ουντίνε Φον Μπλότνιτς εδώ στο Κοινοβούλιο όταν ήμουν συνεργάτη της τότε, είχα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις του Τσερνοβίλ. Και ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα μετά από το δυστύχημα του Τσερνοβίλ ήταν ακριβώς η αδιαφάνεια, η έλλειψη δυνατότητας ευρέως δημοκρατικού ελέγχου. Και μου φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτή τη στιγμή α, επιχειρηματολογούμε αμυντικά και δεν θα πρέπει να ακολουθούμε εδώ την συνθήκη Ευρετόμ αλλά την προστασία των πολιτών βάσει κανόνων ε, των ευρωπαϊκών συνθήκων για να έχουμε πλήρη έλεγχο και πλήρη λόγο σε αυτά. Και θέλω να πω προς τον κύριο Μπαρνιέ, ο οποίος προέρχεται από την Γαλλία, να φροντίσει κάτι να αλλάξει στη Γαλλία γιατί στη Γαλλία τότε δόθηκε εντύπωση ότι τα ραδιενεργά σύννεφα περνάγανε γύρω γύρω από τη Γαλλία και αυτό ήταν πραγματικά ντροπή. Εγώ όπως και η κυρία Χολ θα ήθελα να προτείνω να προσανατολιστούμε ε, στον κανονισμό των ΙΠΑ ε, πολύ συντηρητικό πρακτική προσέγγιση, δηλαδή όχι οριακές τιμές για ενήλικες και παιδιά, για ισχυρούς και για ανίσχυρους, αλλά να προσανατολιστούμε συντηρητικά σε αυτό που μπορούν να αντέξουν τα παιδιά. Πολύ συντηρητικά. η συστάση των ΗΠΑ είναι ένα δέκατο αυτών που αυτή τη στιγμή συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ε, Ευρατόμ. Θα έπρεπε να με ακολουθήσετε και εμένα και κυρία Χολ εδώ. Ευχαριστώ κυρία Χάμψ, εξ ονόματος της ΚΑΕΦΑΟΕΛ, η συνάδελφος Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ αρχίζοντας ε, όπως και οι συνάδελφοι να πω ότι όταν μιλάμε για ραδιενεργό επιμόλυνση των τροφίμων να συζητούμε για ένα θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Ε, επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων ραδιενεργούς μόλυνσης ε, συνδέονται με τις επιπτώσεις επί της δημόσιας υγείας. Αριθμός ε, κρουσμάτων καρκίνου, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μια νομική βάση που να θέτει στον πυρήνα του προβλήματος τη δημόσια υγεία. Οπότε γνωρίζουμε την κατάσταση όχι μόνο λόγω του Τσέρνομπιλ, αλλά και για άλλες περιπτώσεις το Τσέρνομπιλ μας έδειξε το μέγεθος ε, αυτού του προβλήματος κατέδειξε πώς μπορεί να επηρεαστεί η καθημερινή ζωή όλων. Δεν αντλήσαμε τα διδάγματά μας. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να καταπολεμήσουμε οποιοδήποτε επικίνδυνο φαινόμενο. Λοιπόν, είναι σαφής η πρόταση, ε, αλλά θα πρέπει, όπως σας είπα, να επιλέξουμε νομική βάση που να επικεντρώνεται στο θέμα της δημόσιας υγεία. Επίσης, υπάρχουν κάποια καταχρηστικά μέτρα που επαφίονται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών Πρέπει να καταργηθεί αυτό. Επίσης, να προβλέψουμε μια πιο διαφανή, μια πιο δημοκρατική διαδικασία λήψη αποφάσεων για τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τώρα. Δεν μπορούμε να ε, ε, μένουμε σε αυτά τα όρια τους πλέον ευπαθείς ε, ε, πολίτες ε, και μόνο. Την υγεία όλων πρέπει να προστατεύσουμε και πρόκειται για για περιπτώσεις, πραγματικές περιπτώσεις θανάτων και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες. Σας ευχαριστούμε τώρα ένα λεπτό από την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, κυρία Ρόσμπαχ. Εγώ πρόεδρε συμφωνώ απόλυτα με αυτή την πρόταση. Όλα τα νέα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να αξιοποιηθούν για να ενημερώσουμε τις τεχνικές ειδικές προδιαγραφές για την προστασία. Έχουμε νέες επιστημονικές δυνατότητες για την προστασία των ζώων και των τροφίμων. Η ραδιενέργεια είναι εξίσου επικίνδυνη στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε προτάσεις σαφείς οι οποίες θα ενισχύουν τους κανόνες μας. Ευχαριστώ κυρία Ρόσμπαχ. Ένα μισή λεπτό, ο συνάδελφος Τσέγκεντη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ουγγαρία έζησε τις επιπτώσεις του πυρηνικού δυστυχήματος ε, τότε με το Τσερνομπίλ ε, και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Και τμήμα της πρόσληψης πρόληψης είναι ότι θα πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά τις ε, πυρηνικές μονάδες που υπάρχουν είναι σημαντικό να τονίσουμε τον ρόλο ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, προσπαθώντας να μειώσουμε την συμμετοχή της ε, πυρηνικής ενέργειας στο μείγμα της ε, ε, ενέργειας. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε βελτίωση της ασφάλειας. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις πτυχές προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζοντας τι είναι καλό και όχι για αυτούς. Όσον αφορά τα... τις επιπτώσεις των ε, δυστυχημάτων αυτών, των ατυχημάτων, θα πρέπει να μειώσουμε τους ε, κινδύνους για τους πολίτες εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις, ε, τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ συνάδελφο γιατί Οι επόμενοι ομιλητές τώρα. Η συνάδελφο Ρωσίκο Βαμπίνοβα δεν έχει έρθει ήδη. Ένα λεπτό λεπτό ο κύριος Μέλτσερ. Το Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις ε, τότε το 86 έπληξαν τις ε, λόγω χώρες αυτές χωρίς να μπορούν να έχουν προετοιμαστεί καθόλου. Η μόλυνση με ακτινοβολία ορισμένων των τροφίμων μπορεί να είναι σημαντική για πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να τη δούμε ούτε να τη μυρίσουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν ε, τα προϊόντα που έχουν μολυνθεί με ακτινοβολία, όπως παραδείγματο χάρη τα βατόμουρα και άλλα φρούτα των δασών, ε, όχι μόνο επιτόπου και σε άλλες χώρες. Χωρίς κανένας να γνωρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος και οι επιπτώσεις και στους ενήλικες και στα παιδιά εμφανίζονται επίσης μετά από δεκαετίες πολλές φορές. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να έχουμε μόνο τρόφιμα και ζωοτροφές που μπορούν πραγματικά να θεωρηθούν ότι είναι τελείως αυλαβείς. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνεται ακτινοβολία ε, οικοθελώς στα τρόφιμα για λόγους διατήρησης κλπ. Και έχει φτάσει πια η στιγμή όχι μόνο να κλείσουν όλες οι πυρηνικές μονάδες αλλά να σταματήσουν και τα πυρηνικά πειράματα για να μπορεί ο καθένας να τρώει τα μανιτάρια που φυτρώνουν στο δάσος του. Um Ευχαριστώ κύριε Μπέλτσερ. Περνάμε στη δεξιά Κασουδιάη τώρα. Ε, στην άλφος Ντάντσιλα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 σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση γενικότερης μόλυσης και να δώσουμε δημοκρατική νομιμότητα σε έναν κανονισμό σημαίνει ότι καθορίζουμε όρια ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και των λαών που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης. Και τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να ελέγχουν το σεβασμό των καθορισμένων επιπέδων στα τρόφιμα και στις γεωτρήσεις αλλά και στις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ευχαριστώ. Για να κλείσουμε τη διαδικασία Καρσδάης, Μέλπος Φεραίρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ένα πυρηνικό ατύχημα ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ραδιολογική εκτάκτου ανάγκη λόγω του, της που έχει και του διασυνοριακού χαρακτήρα απαιτεί ένα συντονισμό προσπαθειών και τη συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματο διαδικασιών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του ατυχήματο για τον πληθυσμό και για το περιβάλλον. Αυτή η ανάγκη συντονισμού συνδέεται με την θέσπιση ανώτατων επιτρεπτών ορίων για την επιμόλυνση τροφίμων και ζωοτροφών. Δεν μπορούμε όμω να δεχτούμε την επιχειρηματολογία ότι για να εξυπηρετήσουμε, λέει, καλύτερα τα συμφέροντα των πολιτών και για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα ατυχήματα θα πρέπει να ε, περιοριστεί το περιθώριο ελιγμών και η παρέμβαση των κρατών μελών. Το αντίθετο, τα κράτη-μέλη τη βασική ευθύνη για την ε, ε, προάσπιση τη δημόσια υγεία των πολιτών του. Γι' αυτό και για άλλου λόγου, σε περιπτώσει εκτάκτου ανάγκη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν με υψηλά επίπεδα προστασία και να καλύψουν όλε τις διαστάσεις του ζητήματος ε, ε, ε, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους, δηλαδή να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Σας ευχαριστούμε. Πέρα της διαδικασίας του ΚΑΤΣΕΔΙΑΗ και τώρα ο Επίτροπος Μπαρνιέ έχει το λόγο παρακαλώ. Merci, ως πολιτικός και ως πολίτης αυτό που μπορώ να πω. Μα θυμήσατε κυρία Άρμς ότι είμαι Μα δεν φταίει μόνο αυτό. Αυτά είναι θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ όταν ήμουν Υπουργός περιβάλλοντος της Γαλλικής Δημοκρατίας ασχολήθηκα με τη ρήπανση των εδαφών 93-94 με το, Τσερνοβίλ. Όταν πήγα δε στην Ουκρανία, στο Τριπίρτ, μια πόλη φάντασμα, ε, ε, ε αυτά τα οποία είδα δεν τα ξέχασα. Και ως βουλευτής εγώ, εγώ εργάστηκα για την οικολογική προστασία της Ευρώπης. Συνέταξα και έναν Άτλαντα σχετικά για τους κινδύνους παγκοσμίω. Εκεί όπου η κουλτούρα του κινδύνου δεν υπάρχει. Επίσης ήμουνα και υπουργό Γεωργίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για ασφάλεια, για ανθρώπινη υγεία, προστασία των πολιτών, των καταναλωτών, αλλά και για την υγεία των ζώων. Μα όλα αυτά είναι θέματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω τέτοια προχωρημένη ώρα. Υπάρχει ένταση στους βουλευτές και όπως είπα και στον κύριο Μπελέτ, άκουσα πολύ προσεκτικά και θα αναφέρω στους συναδέλφους μου όλες αυτές τις ανησυχίες που τόσο μόφωνα εκφράσατε. Τώρα αυτό το οποίο θέλω να σας πω και το οποίο με δεσμεύει τώρα και από νομικής πλευράς όπου το σώμα των επιτρόπων βασίζεται αυτά είναι τα επιχειρήματα στα οποία βασίζεται και η Κομισιόν Σώμα και η κύριος Σεύκοβιτς και ο κύριος Σότιγκερ νομικοί όροι που λένε ότι η συνθήκη Ευρατόμ για την προστασία προστα... ε, υπερισχύει της ε, συνθήκης της Ένωσης και ότι αυτές οι διατάξεις γίνονται σεβαστές από τις τρεις από τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτά είναι τα επιχειρήματα που αναφέρει και που προβάλλει η Κομισιόν για να απορρίψει τις τροπολογίες. Αλλά εγώ θα αναφέρω στους συναδέλφους μου όλες τις ανησυχίες που εκφράσατε. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Μπέλεκ. Για ακόμη μία φορά καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Εγώ σέβομαι απόλυτα το άτομό σας, τις ικανότητές σας. Ε, εσείς επαυξήσατε βεβαίως όλα αυτά μιλώντας για την εμπειρία σας ως υπουργό Γεωργίας, την επίσκεψή σας στο Τσερνομπίλ κλπ. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει μία κοινή θέση, ένας αγώνας, ένας κοινό αγώνας, ουσιαστικός αγώνας. Το δικαστήριο μας έδωσε μια ιδιαίτερα ομόφωνη ερμηνεία συμβατή με την ερμηνεία και του νομικού συμβούλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για ευρατόμα, αλλά για δημόσια υγεία, άρα εφαρμοστικό πεδίο Λισαβόνας. Ε, λυπούμε για την ισχυρογνωμοσύνη της Κομισιόν που θεωρεί ότι εγώ, που, που, που, εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι η κωδικοποίηση θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αν υπάρξει ένα δυστύχημα ένα ε, ραδιενεργό επεισόδιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από θεσμικής πλευράς εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε τους ισχύοντες κανόνες που σήμερα είναι ανεπαρκείς. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να με ακούσετε. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν πότε θα μας παρουσιάσει την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων για την δημόσια υγεία και τη διατροφή στην δεκαετία του 80 κύριε Επίτροπε όταν εσείς επισκεπτόσασταν το Τσερνομπίλ είχε συνταχθεί ένας νόμος με μία ρήτρα αναθεώρησης. Πότε λοιπόν θα έρθει αυτή η αναθεώρηση? Σας ευχαριστώ κύριε Μπελέτ. Ε, Ολοκληρώνεται την εξέλιξη του θέματος αυτού. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12.